προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ζητούμε ένα κοινό καταστατικό για τι αλληλασφαλιστικέ εταιρείε, του συνεταιρισμού και τα ιδρύματα. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Προχωρώ τώρα στι ψηφοφορίε. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την, πρόταση, την ψηφοφορία για δύο προτάσει ψηφίσματο για τον Ουγγρικό νόμο για τη Μέσα Μαζική Ενημέρωση. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν την ψηφοφορία που προβλέπετε για το ψήφισμα για τα ΜΜΕ στην Ουγγαρία, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στις τελευταίες εξελίξεις της κατάστασης και να κάνω μία συγκεκριμένη πρόταση. Πριν από τέσσερις μέρες, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ε, πέρασε τις ε, τροποποίησεις, όλες τις τροποποίησεις που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά την αρνητική ψήφο των ε, σοσιαλιστικών και πράσινων βουλευτών της Ουγγαρίας. Η Επίτροπος Κρούς ήταν παρούσα και είπε ότι ο τροποποιημένος νόμος ήταν σύμμορφος με το ευρωπαϊκό δίκαιο και κυρίως με την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το ψήφισμα των αριστερών που, που υποβάλλεται στην ψηφοφορία αγνοεί αυτά τα γεγονότα. Το κείμενο είναι ακριβώς το ίδιο με το κείμενο που είχαμε πριν από τρεις εβδομάδες και καθόλου δεν αναφέρει την ψήφο του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Διερωτώ με, ζούμε στην πραγματικότητα ή σε κάποιο φανταστικό κόσμο. Ε, αυτό το ψήφισμα είναι κατά του Ουγγρικού Κοινοβουλίου ή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν έχει τίποτα να πει εναντίον του νόμου αυτού. Ζητώ. Ζητώ από τον πρόεδρο των φιλελεύθερων να δείξει εμπιστοσύνη στην Επίτροπο, Επίτροπο και τον ρωτώ, της έχει εμπιστοσύνη ή όχι. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα χάνε την αξιοπιστία του εάν υιοθετούσε αυτό το κείμενο το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας. Θα πρέπει να ρυθμίζουμε εδώ τους εθνικούς πολιτικούς λογαριασμούς. Αυτό θέλετε. Σε αυτό θα πρέπει να μετασχηματιστούμε. Και σε αυτές τις ε, συνθήκες εμείς αποσύρουμε το κείμενό μας, το κείμενο πρότασης από πλευρά ΣΕΛ και ζητούμε και οι υπόλοιπες ομάδες να κάνουν το ίδιο πράγμα. Είναι θέμα αξιοπιστίας του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, e, e, Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρότασή σας είναι πολύ σαφής. Η ομάδα του ΕΛΚΑ αποσύρει το κείμενο πρότασης ψηφίσματος. Παραμένει μόνο ε, ένα κείμενο που έχουν παρουσιάσει πολλές ε, πολιτικές ε, ομάδες και θα ήθελα οι ομάδες οι οποίες εκπροσωπούνται να πάρουν το λόγο και να εκφραστούν για το σημείο αυτό. Ο κύριο Φάμποντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριο ε, Ντόλ ε, παραπέμπει σε ρεαλισμό και πραγματικότητα. Όντω, είναι πραγματικότητα ότι η Ουγγρική κυβέρνηση τροποποίησε το σχετικό νόμο και καλώ έπραξε. Γιατί θα υπενθυμίσω τη συζήτηση στην οποία και εσεί, κύριε Ντόλ, είχατε πει ότι όλα καλά σε αυτό το νόμο και δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί τίποτα την προηγούμενη φορά. Δεύτερον, όμως η πραγματικότητα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μπορείτε να το διαβάσετε και εσεί στο κείμενο είναι ότι ο ίδιος ο εκπρόσωπος του πολίτη για τα μέσα μαζική ενημέρωση λέει ότι δεν αρκούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και η Επιτροπή αυτό λέει, η τροποποίηση των νόμων δεν επαρκούν. Αυτό είναι η πραγματικότητα κύριε Ντόλ, κύριε συνάδελφε. Στην ομάδα συζητήσαμε υπό δική μου προεδρία χθε διεξοδικά όλε αυτέ τι τροποποιήσει στην ομοθεσία τη Ουγγαρία και επίση είπαμε ότι είναι και ε, με βάση τα όσα μας λέει ο Επίτροπος του Πολίτη, ο πρόσωπος του Πολίτη για τα μέσα και ενημέρωση, αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ανεπαρκής ελλειπείς αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Και εμείς κύριε Λάγκεν, κύριοι συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Αν εσεί συνθηκολογείτε είναι δική σας υπόθεση. Η ελευθερία του τύπου είναι για μας αλληλένδετη αξία και αρχή μέσα σε μια δημοκρατία. Θέλουμε δημοκρατία, θέλουμε ελευθεροτυπία, ελευθερία του τύπου και γι' αυτό ζητούμε να γίνει ψηφοφορία σήμερα. Για να ξέρουν όλοι ότι, εσύ, ότι ε, εμείς αγωνιζόμαστε και όχι εσείς για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την ελευθερία του τύπου στην Ουγγαρία και παντού. Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι υπόλοιπε τέσσερι πολιτικέ ομάδε δεν αποσύρουν την πρόταση ψηφίσματό του. Επομένω, μπορούμε να σταματήσουμε τη συζήτηση και να περάσουμε στην ψηφοφορία. Οι φιλελεύθεροι θα ήθελαν επίση να πάρουν το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έγινε αναφορά στην ομάδα μου, συγκεκριμένα. Και θα ήθελα να πω ότι ναι, έχουμε εμπιστοσύνη στην, ε, ε, στις προσπάθειες και το έργο της Επιτρόπου Κρούς που έχει αποδείξει ήδη την αξία της. Ε, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε τίποτε άλλο να πράξει άλλωστε στην υπόθεση αυτή. Πιστεύω το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, πραγματικότητα είναι αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Σβόμποντα μόλις τώρα και Σα... και ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης μας λένε ότι δεν επαρκούν αυτές οι τροποποίησεις και δεν είναι ουσιώδεις τροποποίησεις στις οποίες ε, προέβη η κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Έχω μιλήσει με τους συναδέλφους του Ούγγρους ε, και μας έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν επαρκούν όλα αυτά. Για την ε, ομάδα των φιλελευθέρων λοιπόν θα ήθελα να πω ότι δεν αποσύρεται η πρόταση ψηφίσματος και ότι ζητούμε να γίνει ψηφοφορία. Ε, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία της προτάσεως ψηφίσματος τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Φέτο την πρόταση ψηφίσματος σε ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας.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 Um não está refletido na resolução. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα ζήτημα που δεν αναφέρεται στο ψήφισμα για τη Λιβύη, για τις κοινωνικές χώρες του Νότου. Θα ήθελα να με στηρίξετε και να εκφράσουμε όλοι μαζί την αγανάκτησή μας αλλά και την ανησυχία μας. Τι εννοώ. Τι έγινε σε αυτούς τους δημοσιογράφους του BBC οι οποίοι κρατήθηκαν παρανόμως και βασανίστηκαν και μάλιστα μέχρι και σε αυτό το βασανιστήριο ε, του ε, Ιωνί θανάτου υποβλήθηκαν. Δεν είναι ανθρώπινες συνθήκες αυτές. Ε, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν ελεύθερα τη δουλειά τους στη Λιβύη. Είναι μια πολύ σημαντική πτυχή αυτή, την οποία νομίζω ότι θα πρέπει να θέσει ε, σαφώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να στείλει έτσι ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο. Εκφράζουμε την αγανάκτηση και την ανησυχία μας. Ο Πρόεδρος, ε, απευθύνομαι στην κυρία Γκόμες. Έχετε μια συγκεκριμένη τρόπο, για να μας ε, προτείνετε, διότι Μόνο γενικές ε, προτάσεις μπορούμε να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Η κυρία Γκόμες, νομίζω ότι η ομάδα των φιλελευθέρων, όπω συμφωνήσαμε, θα καταθέσουν με προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχει, με τα χαράς να σας κάνω εγώ μια πρόταση. Παν Πολύ, πολύ καλά. Ο κύριος Καμίνσκι θέλει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε, είδαμε και την ανακοίνωση, είπατε ότι εγκρίθηκε το ψήφισμα για την Ουγγαρία, αλλά στην οθόνη μου δεν είδα εγώ το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δικαιούμεθα να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ωραία. Θα σας πω λοιπόν 316 ήταν οι ψήφοι υπέρ, 264 ήταν οι αντίθετες ψήφοι και υπήρχαν και 33 αποχές. Ευχαριστώ. Chairman, I would like to remind the House. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επενθυμίσω ε, στο σώμα ότι εφαρμόζουμε διπλά ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά ε, το νόμο για τα ογκρικά μέσα. έγιναν εξελίξεις αυτές τη Δευτέρα, δεν ελαμφέρουμε τίποτε στο ψήφισμα, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα της Λιβύης θέλετε να αναφέρουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάλογα με το θέμα. Ε, Αγαπητοί Παρακαλώ τώρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία τη σχετική με τις προτάσεις ψηφίσματος από πέντε πολιτικές ομάδες για την Λιβύη. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ε, ε, ονομαστική ψηφοφορία στην παράγραφο υπαριθμών 10, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η ομάδα των φιλελευθέρων θέλει να καταθέσει μια προφορική τροπολογία στην υπαριθμόν 11 παράγραφο. Ο κύριος ε, Φερχόφστατ, παρακαλώ εκ μέρου ε, των Προέδρων όλων των πολιτικών ομάδων και των Πεστών Συντονιστών καταθέτω την πρόταση, Προέδρε, διότι εχθέ έγινε μια συζήτηση από την οποία προέκυψε ο γενικό αίσθημα ότι θέλουμε να ενισχυθεί το κείμενο στην παράγραφο 11, να καταστεί πιο σαφέ δηλαδή. Η προφορική τροπολογία την οποία καταθέτουμε έχει ω εξή. Καλή την ανώτατη αρχή να αναπτύξει σχέσεις με την προσωρινή ε, μεταβατική, ε, με το προσωρινό μεταβατικό εθνικό συμβούλιο και να ξεκινήσει μια διαδικασία ώστε να αναγνωριστούν επισήμως. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ολόκληρη η τροπολογία χρειάζεται. Ναι, καλή την υπατή εκπρόσωπο να αναπτύξει σχέσεις με, την, ε, με το προσωρινό Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο και να ξεκινήσει τη διαδικασία για την μετατροπή του σε επισήμου έτσι ώστε να διευκολύνει τη μετάβαση στη δημοκρατία, την εξασφάλιση εμπλοκή ευρύτερου του φάσματο των εκπροσώπων τη κοινωνία τη Λιβύη και την α, ε, ανάπτυξη πρωτοβουλία και από πλευρά των γυναικών και των ε, μειονοτήτων έτσι ώστε να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, να την υποστηρίξει για την, να υποστηρίξει αυτές τις μεταβολές, απελευθερωμένες περιοχές και να βοηθήσει τον πληθυσμό προσφέροντας τις απαραίτητες ανθρωπιστικές ε, βοήθειες. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε λοιπόν. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Μπορούμε να περάσουμε σε ψηφοφορία λοιπόν. Ποιο είναι υπέρ αυτή της τροπολογίας. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Παράγραφο 23. Χωριστή ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ψηφίζουμε το σύνολο την πρόταση ψηφίσματος, κοινού ψηφίσματος, με ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Θέλετε να σας κοινοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία. 584 υπέρ, 18 κατά. Τεράστια πλειοψηφία. Είναι σπάνιο αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Τώρα, ψηφίζουμε την έκθεση του κυρίου Μπέλντερ για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράν. Εξετάζουμε την πρόταση ψηφίσματος. Ψηφίζουμε την τροπολογία 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 2 με χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ο κύριος Μπέλντερ θέλει να προτείνει μια προφορική τροπολογία που αφορά την νέα παράγραφο 6. Κύριε Μπέλντερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, με πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και με συμφωνία με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες θα ήθελα την εξή ε, με, τροπολογία μετά την ε, τροπολογία 6, την 6α. Ε, καταδικάζει την ε, παράνομη κράτηση των αρχηγών της αντιπολίτευσης της, του Ιράν, τον κύριο Μουσάβη και τον κύριο Καρούμπη, μαζί με τις γυναίκες τους από τις Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και ζητάει την πάρα αυτή απελευθέρωσή τους. Τονίζει ότι η κράτηση αυτή έγινε κατά παράβαση του Ιρανικού δικαίου. Καταδικάζει τη στάση των Ιρανικών αρχών απέναντι στην αντιπολίτευση που ασκεί το, το νόμιμο δικαίωμά της και δηλώνει ότι είναι αλληλέγγυα με τον Ιρανικό λαό ε, στις δημοκρατικές του προσδοκίες. Ε, θλίβεται για την υποκρισία το, της Ιρανικής κυβέρνησης ε, που ασκούν υπερβολική βία, εκφοβισμό ε, και αυθαίρετες συλλήψεις εναντίον ε, κάποιων φιλιρινικών διαδηλωτών ε, που εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους με τον Αιγυπτιακό λαό στις 14 Φεβρουαρίου. Είναι κανένα που αντιτίθεται σε αυτή την προφορική τροπολογία πριν ψηφίσουμε. Όχι, ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. Ψηφίζουμε την ε, τροπολογία 2 με χωριστή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 37. Σε τμήματα. πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Παράγραφος 39. Χωριστή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Παράγραφος 40. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 3. Χωριστή ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Α, θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 281 ψήφι υπέρ, 315 κατά. Παράγραφος 53 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, άποχες, υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα, προ, υπέρ, κατά, άποχες, υιοθετείτε. Τροπολογία υπαριθμών 1. Χωριστή ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Υιοθετείτε. Πολύ ωραία. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Χωριστή ψηφοφορία. Ένα ψηφοφορία ψήφισαν όλοι. Πέρας. Υιοθετείτε. Το εκτιμώντας K σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Άποχες, υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Άποχες, υιοθετείτε. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Άποχες, υιοθετείτε. Θεολογική σκέψη εκτιμώντα L, Χωρί την ψηφοφορία, υπέρ. Κατά. Αποχές, υιοθετείτε. Το εκτιμώντα N, η κυρία Ιμπρισάγετς θέλει να ε, προτείνει προφορική τροπολογία στο εκτιμώντας n. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. θέλω να κάνω μια προφορική πρόταση τροπολογίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε για την ε, απλή λέξη και. End. Δεν θέλω να διαγραφεί αυτό από το κείμενο. Και θα σας εξηγήσω γιατί λέμε ότι υπάρχει μια σημαντική βάθη στη σχέση μεταξύ Ιράν και Τουρκίας. Και, και αυτό το και θέλω διαγραφή, δεδομένου ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τους ε, του επισήμους και εμεί, στη Συρία, τη Χεσμολάχ, τη, τη Χαμάς αλλά και τους αδελφούς μουσουλμάνους για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Εδώ λοιπόν το και θέλουμε να διαγραφεί γιατί θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να συζευχθεί αυτή η βελτίωση εμβάθυνσης εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Ιράν με την Χεσμολάχ και την ε, Χαμά. Ποιο αντιτίθεται σε αυτή την προφορική τροπολογία. Κανεί. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία, την προφορική που αφορά το εκτιμώντα 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ υιοθετείται το εκτιμώντας O, όμικρον, τη ψηφοφορία, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος της αρμόδιας επιτροπής, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τώρα, ψηφίζουμε τις έξι προτάσεις ψηφίσματος για την 16η Σύνοδο του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κυρία Άουταλα, της, η πρόεδρος της Υποεπιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Χάουταλα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια πολύ καλή είδηση. Ο κύριος Χαϊτάμαλ Μαλέχ... Ε, ε, 80 χρονο δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη Συρία έλαβε άφηση και ε, χάρη συγκεκριμένα και απελευθερώθηκε πριν από δύο μέρε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε ότι τελικά ε, κάποιες φορές εφαρμόζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Ο εν λόγω δικηγόρο πραγματικά ε, έχει αγωνιστεί και θα συνεχίσει να αγωνίσει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία. Ευχαριστώ. Dziękuję pani za tę wypowiedź. Na pewno wszystkich. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία κυρία Χάουταλα. Είναι πολύ ενθαρρυντική και θα μας οθήσει να συνεχίσουμε τη δράση μας. Προχωράμε λοιπόν τώρα στην πρόταση, στις προτάσεις ψηφίσματος. Ε, αυτές πρώτα απ' όλα παράγραφος 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 8 τροπολογία 2 ψήφι υπέρ. Κατά θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Η τροπολογία 2 απορρίπτεται. Επομένως ψηφίζουμε την παράγραφο 19 με χωριστή ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ήταν η παράγραφος 8. Παράγραφος 19. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 39. Χωριστή ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα το ελέγξω ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης κοινού ψηφίσματος. Ναι, παρακαλώ διαδικαστικό. Θέλω να σας επισημάνω ότι όταν θέσατε σε ψηφοφορία την παράγραφο 8, το αρχικό κείμενο, όλοι ακούσαμε άλλο, άλλον αριθμό, ε, οπότε θα ήθελα να επαναλάβετε την ψηφοφορία. Δεν έγινε κατανοητό για ποια παράγραφο ψηφίζαμε. Λυπούμε. Ε, θα ε, θέσω ε, πάλι σε ψήφιση όλο το σύνολο του ψήφιματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι δεκτό με μεγάλη πλειοψηφία το κοινό ψήφισμα. Κύριε Λαντσμπέργκης, θέλετε να λάβετε το λόγο. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Ευχαριστώ όλες και όλους. Thank you, Diana. No, thank you. Have a good weekend. Thank you. Before we move to the explanations of votes, I have a point of order. Πριν προχωρήσουμε, έχει στήσει η κυρία Χόλ μία, ε, ένα διδικαστικό ως προς τις γραπτές δηλώσεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζητώ μόνο να έχω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους 400 συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες που συνυπέγραψαν την γραπτή δήλωση παριθμών 81 αλλά και το προσωπικό του γραφείου μου που με στήριξε με σκληρή δουλειά και τις υπηρεσίες των γραπτών δηλώσεων για την υποστήριξή τους. Πάνω απ' όλα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι αγωνίστηκαν στην εκστρατεία για αυτή τη γραπτή δήλωση που κατέστησαν δυνατή αυτό το αποτέλεσμα. Και αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια που είμαι και εγώ μέλος ενός κοινοβουλίου το οποίο, χάρη στο οποίο μπορεί ο κοινό πολίτης να προσφέρει, να προτείνει τα επιχειρήματά του, να τον ακούσει ο βουλευτής και να πιστεί από αυτά τα επιχειρήματα. Αυτή είναι η δημοκρατία η πεμπτουσία της δημοκρατίας αποδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί μακριά από τον πολίτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χόλο. Επεξηγήσεις ψήφων τώρα. Καταρχάς για το νόμο περί μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ουγγαρία, η κυρία Μπένοβα.